Ο κύριο Βαλέσα, για παράδειγμα, ευχαριστώ όλου του άλλου συναδέλφους. Εδώ διακόπτεται η συνεδρία και επαναλαμβάνεται στι 3 του μεσημέρι.